θα, ξεκινήσουμε τη συνεδρία μας. Hello. je commence par vous rapporter. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω ε, καλ... ζητώντας την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω τα, ποια είναι τα αποτελέσματα από τη συνεδρίαση των συντονιστών προχθές. Διαδικασία επιτροπολογίας. Έχουμε τις επιστολές 14 και 15, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχόλια για τα θέματα αυτά. Δεν προέκυψαν ιδιαίτερα ζητήματα ως προς το 14 και 15. Τώρα, ως προς το αεροπορικό πακέτο, οι τρεις εκθέσεις θα ψηφιστούν στην Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου, ούτως ώστε να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση του κυρίου Ουτζίας ε, θα είναι το Σεπτέμβριο κάποια στιγμή. Τώρα, ως προς τον προϋπολογισμό 2013 και τα πιλωτικά σχέδια, η απόφαση είναι ότι θα προτείνουμε να συνεχιστούν οι τρεις προπαρασκευαστικές δράσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί και να μην υποβληθούν νέες προτάσεις. δεδομένου του περιορισμένου ε, προϋπολογισμού που διατίθεται. Ως προς την εβδομάδα της κινητικότητας, ο πρόεδρος της Επιτροπής θα συντάξει μια επιστολή, την οποία θα απευθύνει στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, του ώστε να ζητήσει άδεια να οργανωθεί μια μίνι ακρόαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταφορών το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Τίσντέιλ, διευθυντής της αξιολόγησης αντικτύπου, διαχειριστής αυτού του θέματος και του κόστους της μη Ευρώπης αξιολόγηση του αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή προστιθέμενης Αξία. Απόφαση είναι ότι οι συντονιστέ σημειώνουν όλη αυτή τη δουλειά που έχει ξεκινήσει προ την καινούργια αυτή κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν για του συντονιστέ, Έχετε ερωτήσει, Εάν όχι, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να καθίσετε όμως και να υπάρξει ησυχία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ για περισσότερη ησυχία. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας σας. Να κάνουμε μια δοκιμή παρακαλώ, για να δούμε ότι δουλεύει. Για να επαληθεύσουμε ότι ίσως ως συνήθως τα μέλη του ΕΛΚΑ είναι υπεράριθμα. Άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμή. Κάποιες ψήφοι λείπουν ακόμα. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Τρεις λείπουν. Λοιπόν. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Ποιος δεν ψήφισε. λοιπόν πέρα της ψηφοφορίας. Λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Καλώς. 42 ψήφισαν. Και εκπροσωπούνται κανονικά όλες οι πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε λοιπόν. Τέσσερις είναι οι ψηφοφορίες σήμερα μακρύς ο κατάλογος, περίπλοκος κάπως. Θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση και να προχωρήσουμε με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο και εύρυθμο τρόπο. Αναδιατύπωση του πρώτου πακέτου για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Είστε έτοιμοι. Τροπολογία 1. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. εγκρίνεται αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 αποσύρεται. Τροπολογία 119. Η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αυτή αποσύρεται. Συμβιβαστική λύση Παριθμών 1. Η εισηγήτρια είναι υπέρ προφανώς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία. Οι 120 και οι 122 ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ, η συγγήτρια είναι υπέρ. Όχι, καταπίπτουν, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 5. Όχι, πάμε στην τροπολογία 121. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 5. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. Η 6. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. υπέρ, κατά, αποχές. Κυρία Σνάισερ. Ντομινίκ, δεν χρειάζεται να μας λες ε, η συγκήτρια είναι υπέρ, κατά, όλοι ξέρουμε τι θέλει, έχουμε μια λίστα και έχουμε και πολλές ψηφοφορίες μπροστά μας. Μια πρόταση κάνω απλώς. Όχι. alors nous Καλώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία χωρίς να μιλάω ε, για την ε, άποψη του εισηγητή, της εισηγητρίας. Τροπολογία υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές. Κατά εγκρίνεται. Οι 124 και οι 125 δεν είναι παραδεκτές. Η συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική λύση παριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 126. Το δεύτερο τμήμα κατά προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά θα το επαληθεύσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεκατρία. Προσθήκη επίσης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 5. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 14 και 127 καταπίπτουν. 128 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Όχι, καταπίπτει 16, με συγχωρείτε. Η 17. Ψηφίζουμε τη 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 129 καταπίπτει, η 18 αποσύρεται, ε, συμβαστική τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 130 και οι 19 καταπίπτουν, Οι 131 δεν ήταν παραδεκτή, συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, καταπίπτει, Οι 132, με προφορική τροπολογία. Διαγράφονται οι λέξεις των ρυθμιστικών αρχών Υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Με με την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. και 133 καταπίπτουν. Πρόταση προφορικής τροπολογίας εδώ. Προφορική τροπολογία που την ε, αποφασίσαμε χτε όλες οι ομάδες μαζί. Η τελευταία πρόταση να μην λέει εντός 6 εβδομάδων από τη λήψη των σχετικών πληροφοριών, αλλά εντός 10 εβδομάδων από τη λήψη της αίτηση για να μπορούμε να επεκτείνουμε το χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, δέχεστε την προφορική τροπολογία. Καλώς. 134 λοιπόν ψηφίζουμε μαζί με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχή, αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 22 καταπίπτει. 135 ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία πάλι να διαγραφούν οι λέξεις των ρυθμιστικών αρχών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 πίτη. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 24 καταπίπτει. Η 25. Μαζί με την προφορική τροπολογία, την ίδια, να διαγραφούν οι λέξεις των ρυθμιστικών αρχών, ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές. Κατά. Εγκρίνεται. 138 και 27. Οι τροπολογίες αυτές πίπτουν. Οι 137 όμως όχι. Όχι, και η 137 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στην 28. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Από το requests by ετείται ότι και ολοκληρώνεται στο railway σιδηρόδρομος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεν ξέρω, πονάει το χέρι σας και δεν έχετε ψηφίσει ως χειρός. Ξεκινούμε λοιπόν το τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Ματιέ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Έχω μια ερώτηση για την 137, με συγχωρείτε με την συμβαστική τροπολογία 8 που εγκρίναμε, καταπίπτει 138 συνεπώ. αλλά όχι 137 και την 137 δεν την ψηφίσαμε. Νομίζω ότι είναι τυπογραφικό λάθος. δεν είναι 138 και 138, δύο φορές 138 που βλέπετε στο κείμενο. Θα πρέπει να είναι μία φορά 137 και μία φορά 138. Εξού και έχει όντως καταπέψει 137. Καλώ ευχαριστώ. Πάμε στη 28, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 28. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 139 καταπίπτει. Η 29 αποσύρεται. 141 και 142. Είναι ίδιες οι τροπολογίες σε αυτές. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30 καταπίπτει. Την 140 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Αυτή αποσύρεται. 143. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 32 αποσύρεται. Η 144. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 33 καταπίπτει. Η 145. Ε, ψηφίζουμε αυτήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει. 146 και 147 ψηφίζουμε μαζί για την ίδια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Οι 147 και 36 της εισηγήτριας είναι ίδιες, τις ψηφίζουμε μαζί, υπέρ. Αποχές, κατά, εγκρίνονται. Αποσύρεται 37, 148, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 38 καταπίπτει. Αποσύρεται η 39, 149 της εισηγήτριας και 150 του κυρίου Τσίλε. Είναι ίδιες, τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνονται. Η 40 της εισηγήτριας, ποιος είναι υπέρ, Όχι, με συγχωρείτε, η 40 καταπίπτει μαζί με τις προηγούμενες. Η 151. Ποιος είναι υπέρ της 151. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 43 καταπίπτει. 152 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 44 καταπίπτει. 45 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά. Εγκρίνεται. 49 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50. Αποσύρεται. 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. «155 και 51 καταπίπτουν. 156 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 52 καταπίπτει. Η 53 και οι 157 αποσύρονται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 10 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 και 54. Οι τροπολογίες αυτές καταπίπτουν. Η 55 αποσύρεται. 56 της εισηγήτριας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία υπεριθμών 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 και 58 καταπίπτουν οι τροπολογίες αυτές. Συμβιβαστική το υπαριθμών 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160, 59, 186, 107 καταπίπτουν. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 62 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64, 65, 66, 67 αποσύρονται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. «68 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 και 71 αποσύρονται. 161 της κυρίας Βουίλς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Η ρυθμιστική αρχή μέχρι την παρούσα οδηγία. Αυτό το τμήμα του κειμένου ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Τα κράτη-μέλη μέχρι ότου υιοθετώντα τι αποφάσει. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 163 της κυρίας Wills. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 καταπίπτει. 73 αποσύρεται. 165 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 76 καταπίπτει. Η 74 αποσύρεται. 75 υπέρ. Κα... Αποχές. Κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μάικλ, παρακαλώ. Η επόμενη 167 εκεί πέρα λέμε πάλι το ίδιο. Εντός 6 εβδομάδων να αλλάξει και να γίνει εντός 10 ε, εβδομάδων από την ε, λήψη της ε, καταγγελίας. Συμφωνήσαμε χτες όλοι οι συντονιστές. 167 Qui vote contre Qui s'abstient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 Τροπολογία 101 καταπίπτει, συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 102 καταπίπτει, 103 της ηγέτρες πίνει υπέρ. Κατά. Κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 104 της ηγέτρες υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 184 της κυρίας Βίλς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185 της κυρίας Βίλς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105 και 106 αποσύρονται. Τροπολογία 109 έχει επίσης αποσυρθεί. Τροπολογία 109 της κυρίας Βίλς. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 110 έχει αποσυρθεί. Η 111 της κυρίας Βίλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 112 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 113 δεν γίνεται αποδεκτή η ε, 114 παρακαλώ. αποχή δεκτή. 115 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 116 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 28 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117 καταπίπτει συμβαστική υπαριθμών 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέλος η 118 καταπίπτει. Καταλήγουμε στην τελική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στην κυρία Σερακανή. 20... 35 ε, υπέρ 6 κατά μία αποχή. Νομίζω ότι στηρίζεται με αρκετά ισχυρή θέση. Ε, και πιστεύω ότι θα έρθουμε στην εντολή των διαπραγματεύσεων αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, περνούμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Η ε, ψηφοφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι η έκθεση του κυρίου Τάτορένα. Όχι, συγγνώμη, του κυρίου Κολιτσέκ. Κύριε Κολιτσέκ, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το επισημάνατε. Έκανα ένα μικρό λάθος εδώ, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, περνούμε τώρα στην ψηφοφορία αυτή. Αρχίζουμε με την τροπολογία υπαριθμών 21 της κυρίας Τικάου. 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Τροπολογία 22. Βλάστο, Ντεβέρα και Νταντάμ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 του κυρίου Ταταρέλα και Φιντάντζα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 24 της κυρίας Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 25. Βλάστο Ντεβεράκ Νταντάμ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Ποιος είναι κατά. Αποχές δεκτή. Ο κύριος ε, Κατσιάν κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με τη δημόσια τάξη. Η 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Φτάνουμε στη συμβαστική υπαριθμών 1. Ποιοι είναι υπέρ κατά άποχες δεκτή. Οι 26 και 29 και 4 και 28 καταπίπτουν και φτάνουμε στην 30 του κυρίου Πίρκερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. 31. Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32. Φιντάντσα, Ντανέλη, Σούτζι, Εσταταρέλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 της κυρίας Τικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 του κυρίου Λαζάκη, Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 35. Φιντάντσα, Πύρ και Ντανέλη Σουτζάζη Τεταρέλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36. Ούτζιας. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37. Τιτσά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 38 πάλι Τικάου, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 και 40 της κυρίας Τικάου, unblock, ποιοι είναι υπέρ, κατά, άποχες. Προτείνω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 5 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αμπλοκ τροπολογία 41 και 42 του κύριου Κράμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές πάντα μπλοκ, τροπολογιες 43 43-44 του κυρίου Κράμερ υπέρ κατά αποχές δεκτές οι δύο τροπολογίες τροπολογίες 45 και 46 και πάλι από κοινού ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές Πάντα unblock. οι ε, <laughs> τροπολογίες Κράμερ πηγαίνουν 2-2. 47 και 48 του κύριου Κράμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. <laughs> Πάντα του κυρίου Κράμερ. Πάντα ζευγάρια οι τροπολογίε 49 49-50 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές Άλλο ζευγάρι, 51 και 52 του κυρίου Κράμερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 53 και 54 Κράμερ. Πάντα του κυρίου Κράμερ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Βλάστο Βεράκ Νταντάν. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1, 10, 11, 7, 8, 9 καταπίπτουν ε, σύμφωνα με τη συμβαστική. Τροπολογία 12. Higgins υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Ντεβεράκ βλάστο νταντά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 14. Βεράκ βλάστο Ταντάν. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 κράμερ υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με 21 υπέρ και 19 κατά. Τροπολογία 16 του κυρίου Βλαζάκ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17. Ντεβεράκ βλάστο νταντάν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. Οι 18, 2 και 19 καταπίπτουν. Οι 20 καταπίπτει όπως επίσης και η 3 και περνούμε τώρα στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία Ωραία, έχουμε ακόμα ένα λίγο Υπομονή ακόμα και τελειώνουμε. Πέρα της ψηφοφορία λοιπόν λοιπόν, 37 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε ε, Κολιτσέκ. Εξαιρετική ψηφοφορία. Και ε, πριν ε, μάλλον τώρα περνούμε στην, έκθεση της κυρίας Τικάου για τη στρατηγική ε, σχετικά με την περιοχή του Αθλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε μια επικαιροποίηση της ψηφοφορίας και υπήρχαν αρκετά προβλήματα τα οποία εκκρεμούσαν, προτείνω σήμερα να δεχθούμε και να μην δεχθούμε, συγγνώμη, προφορικές τροπολογίες πέραν αυτών οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί σχετικά με την έκθεση. Μιλάμε για τους ταχυγράφους, ε, ταχογράφους. Σας το είπα αυτό εκ των προτέρων, Πρόεδρε. Σας το είπα εκ των προτέρων. Ματιό, θα ήθελα να επαναλάβεις. Να το επαναλάβεις όταν θα χρειαστεί. Ωραία, υπενθυμίζω για να μην κάνετε λάθος τον κατάλογο. Μιλούμε για την περιοχή του Ατλαντικού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε όλοι έτοιμοι Αρχίζουμε με την συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και οι τροπολογίες 1-2 καταπίπτουν. Συμβιβαστική υπαριθμών 2. καταπιπτουν συμβιβαστικη υπαριθμόν Κατά. Αποχές δεκτή. Οι 3, 4, 5 και 6 καταπίπτουν. Τροπολογία υπερθμών 7 της κυρίας Αγιάλα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 8. Δεβεράκ, Βλαστό και Λεμπρόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Οι 9, 10 και 11 καταπίπτουν. Έχουμε τη συμβαστική παριθμών 3 καταρχήν υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άρα λοιπόν οι 9, 10 και 11 καταπίπτουν. Η τροπολογία υπαριθμών 12 με μια προφορική τροπολογία της κυρίας Τεξέρα. Αυτή έχει κατατεθεί κανονικά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, αυτή η προφορική τροπολογία, η 13 τώρα, Τέιλορ, ως προσθήκη, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, τροπολογία 14 Μόλζελ, ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15, Μπιλμπάο. προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 16, τεξέρα, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 17, Ντεβεράκ Βλαστό, Λεμπράν, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή, 18, Μπιλμπάο ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, συμβιβαστική υπαριθμών 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Καταπίπτουν ή καλύπτει η συμβαστική τη 19-20-21, τροπολογία Βιλμπάου υπαριθμών 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι, είναι, ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, πράγματι 16 προς 20 καταπίπτει. Είμαστε στην 23. Μέλτζερ ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Ακριβώς η ίδια πλειοψηφία, άρα απορρίπτεται. Ε, η ίδια αίσθηση απόρριψης. Λοιπόν, τροπολογία υπέρ 24 Μπιλμπάου υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote fermé. Πέρας. 22 υπέρ 18 κατά, δεκτή λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 25, Βλάστο και Ντεβεράκ, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 Μόλζερ, υπέρ κατά απορρίπτεται 26 Μπιλμπάο ως προσθήκη ποιοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 Μπιλμπάο υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 29 Αγιάλα υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Παράγραφος 12 τώρα, τροπολογία υπαριθμών τέξα, είναι προφορική ψηφοφορία που κατατέθηκε ε, υπό μορφή ε, προφορική υπέρ, κατά, αποχές, δέκτη και περνούμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και συγχαίρουμε την κυρία Τρικάου διότι εγκρίθηκε με 37 υπέρ, 3 κατά και 0 αποχές. Είδου λοιπόν. <laughs> Ε, κύριε Γκρός. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Για να μην ε, τα λέμε συνεχώς γαλλικά, θα μιλήσω στα γερμανικά. Το ΕΛΚ ζήτησε αναβολή της ε, ψηφοφορίας γιατί θέλουμε να συντονίσουμε κάποια πράγματα και εσωτερικά και με τις άλλες ομάδες στο σημαντικό αυτό θέμα. Γι' αυτό υποθέτω πως μετά τη σημερινή πλειοψηφία και μέχρι την Ολομέλεια θα καθίσουμε με τις άλλες ομάδες για να επιφέρουμε κάποιες διορθώσεις. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να μην δεχτούμε άλλες ε, προφορικές ε, τροπολογίες ή χωριστές ψηφοφορίες, πλην βεβαίως όσων περιλαμβάνονται ήδη στην ε, λίστα. Δεν είναι θέμα κάποιας ε, επιμονής. Απλά το κείμενο εδώ πέρα, μπορώ να σου το πω, δεν είναι αυτό το οποίο πολλοί συνάδελφοι περίμεναν. Γι' αυτό ακριβώς ε, περιμένουμε πάρα πολλές ε, διορθώσεις. Ευχαριστώ. Δεν έχω σχόλια να κάνω. Υπενθυμίζω ότι η απόφαση για ε, αναβολή της ψηφοφορίας υπήρξε αντικείμενο συζήτησης ευρείας γι' αυτό και καταλήξαμε στη σημερινή ψηφοφορία βεβαίως ε, το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό ε, η τροπολογία ορό θα κατατεθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και με ξεχωριστή ψηφοφορία αυτό προβλέπει ο κανονισμός η κυρία Φώστερ θέλει να λάβει το λόγο παρακαλώ κυρία Φώστερ έχετε το λόγο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί, του, επί της διαδικασίας σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Ρώστερ, πρόκειται για ένα σύνθετο ε, φάκελο που και οι περισσότεροι εξημών θεωρούμε ότι δεν είχαμε επαρκή χρόνο για να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Ε, πολλοί, ε, πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Σαΐτ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, ήδη αναβάλαμε την ψηφοφορία για μία φορά. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρός ότι συνήθως μετά την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή και την Ολομέλεια υπάρχει ε, δυνατότητα για συνάντηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων και αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα. Συνεπώς η ομάδα μου είναι ε, έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι. Ας δούμε πρώτα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και βλέπουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει το αίτημα να μην υπάρχουν ούτε προφορικές ούτε και ξεχωριστές ψηφοφορίες και αυτό προβλέπεται από το κανονισμό και τόσο η συγητής όσο και η σοσιαλιστική ομάδα παραμένουν ανοιχτοί μετά το πέρας της ψηφοφορίας για περαιτέρω συντονισμό. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ να είστε προσεκτικοί αλλά και να επιδείξετε κατανόηση διότι είναι ε, σύνθετο το ζήτημα και πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά. Α, ήδη με ενημερώνουν ότι υπάρχουν λάθη στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε αργά και προσεκτικά. Σας παρακαλώ μη μου πετάξετε ντομάτες. Λοιπόν, αρχίζουμε. Με την τροπολογία υπαριθμών 7 πρόκειται για τροπολογία του εισηγητή τεχνικής φύσεως προφορική κατατέθηκε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνούμε στις συμβαστικές. Ε, Συμβιβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Η συμβιβαστική υπαριθμών 1 εγκρίνεται. Συνεπώς, τροπολογίες 8, 9, 10, 11, 134, 166 και 135 καλύπτονται και περνούμε στην υπαριθμό 136 και 137 που είναι ταυτόσιμες και προτείνουμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Ε, Κοχ και Φέρμπερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Απορριπτώνται. Ε, λοιπόν, έχουμε τις γκρι σελίδες, αφορούν στη συμβαστική 2, διότι το σύνολο των άρθρων ε, στην τροπολογία 136 καλύπτουν. Φτάνουμε λοιπόν τη συμβαστική 2, επί του άρθρου 3. Ε, συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική υπαριθμών 2 εγκρίθηκε. Η 167 αποσύρθηκε. Παραμένουμε στις γκρι σελίδες. πρέπει να το βρω όμως, γιατί έτσι όπως είναι μες, στα, στη μαυρίλα δεν το Α, βρήκαμε την συμβαστική 3 επί του άρθρου 4. Ο κύριος Γκρόσου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι η τροπολογία 184 στο πρώτο μέρος δεν καλύπτεται από τη συμβαστική 3. Τώρα θα ψηφίσουμε ή δεν θα ψηφίσουμε, πρέπει να το γνωρίζουμε. 184, Η 184 δεύτερο μέρος. Δεν υπάρχει τίποτα αντίθετο και ούτε και συμπεριλαμβάνεται όμως τη συμβαστική. Και αισθάνομαι σε θέση μειοψηφία. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ζητείτε να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος της 184. Ωραία. Νομίζω ότι είναι λογικό να το αποδεχτούμε αποδεχθούμε αυτό. Κυρία Τικάου. Κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες με τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Όλοι οι σκιώδες συμφώνησαν, όλοι οι τροπολογίες που καλύπτονται με γκρι χρώμα καλύπτονται από την συμβαστική. Προτείνω λοιπόν να παραμείνουν οι συμβαστικές ως έχουν και αν είναι απαραίτητο βλέπουμε στην Ολομέλεια και συζητάμε με τον κύριο Γκρός αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτό το κομμάτι της τροπολογίας του. Εγώ όμως προτείνω να διατηρήσουμε τις συμβαστικές ως έχουν. Ο πρόεδρος, κοιτάξτε, για να απλοποιήσουμε τα πράγματα έτσι και να ξέρουμε τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να θέσουμε το θέμα υπό την σοφία της ε, πρέπει να δεχθούμε άπαξ απαντός τις θέσεις του εισηγητή. Είτε αυτό που μας λέει ότι όλα καλύπτονται και άρα δεν υπάρχει κανένα αίτημα ή εάν η πλειοψηφία εδώ δεν είναι υπέρ αυτής της άποψης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα σχόλιά του. Να, είμαστε, να επιδείξουμε συνοχή. Ποιοι είναι υπέρ της άποψης ε, του εισηγητή ότι το σύνολο που καλύπτεται από τη συμβαστική δεν μπορεί να διαιρεθεί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. <laughs> Εντάξει, τέλεια. Ωραία λοιπόν, επανέρχομαι στην ψηφοφορία μου. Λοιπόν, συμβιβαστική υπαριθμών 3, αν δεν τα μπέρδεψα, επί του άρθρου 4. Λοιπόν, συμβιβαστική υπαριθμών 3, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Και άρα, περνούμε στην ε, Συμβαστική 4, γιατί πρέπει να βρούμε τις συμβαστικές μέσα στις γκρίμα Λοιπόν, συμβαστική παρισμόν 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άρα τώρα πηγαίνουμε κατευθείαν στη σελίδα 10. Βρίσκεται τη συμβαστική παριθμόν 5 la 5, euh, Συμβαστική υπαριθμόν 5, ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ευχαριστώ. Αμέσως μετά πιο κάτω είναι η συμβαστική υπαριθμόν 6. Il faut les voter. Alors, on va commencer par voter le compromis. Ωραία. Αυτά βρίσκονται στη συμβαστική 6. Ψηφίζουμε καταρχήν τη συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αλλά κάποιες τροπολογίες σχετικά με το άρθρο 16 η 76 η 76 του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία 76 του εισηγητή λοιπόν ποιοι είναι υπέρ Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Il y a manque trois encore, petit petit. Nous avons, il y a manque encore trois, carte qui est revenue. Encore deux petits, petits, petits. Attention, on va fermer. On va fermer, on va. Πέρας της ψηφοφορίας. Oh. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. 19 κατά 18 υπέρ. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11, συμβιβαστική 11, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική. Τροπολογία Υπαριθμό 12. Να κάνουμε εδώ μια διόρθωση. Έχει προσθεθεί κάτι στο κείμενο η πρώτη πρόταση. Αξιολόγηση αντικτύπου για τη σκοπιμότητα και την αξία and merit. Αυτό είναι που προστίθεται. And merit. Όπως τροποποιήθηκε λοιπόν ή όπως διορθώθηκε αν θέλετε ε, Ποιο είναι υπέρ τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμό 12. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλώ. 86 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται, αλλά να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ και 18 κατά. 24 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Όχι 24, 244. Μαζί με την τροπολογία του κυρίου Μπαχ. Τη 2.45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.46 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 91 της εισηγήτριας μαζί με την 271 της κυρίας Σενάλοβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 273 του κυρίου Βαντάλεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 272 του κυρίου Χίγκινς Τον κυρίων Χίγκινς, Λεβρέχτ, Κοχ και φιντάντσα. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτές. Δεκτή η τροπολογία. 2.74 του κυρίου Ούλμερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.75 του κυρίου Ούλμερ υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς αν έχετε την καλοσύνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή η τροπολογία. 93 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 286 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Όχι, με συγχωρείτε, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 17. Αυτή ψηφίζουμε τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 286 της κυρίας Λίχτενμπεργκερ. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Πράγματι εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ 19 κατά. 2.89 του κυρίου Φαντάλεν. Ή μάλλον όχι. Ναι, ναι, πρέπει να την ψηφίσουμε την 289. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα που πάμε. Πάμε στην 333 του κυρίου Καντράουι και της κυρίας Τιτσάου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρία έντεκα. Καταπίπτει νομίζω. Όχι. Ε, το υψηφίζουμε τη 311. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 309 της κυρίας Αγιάλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν έχει και μεγάλη επιτυχία. Απορρίπτεται. 308. Δεν την ψηφίζουμε. Επομένως είσαστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Καλώς. Ψηφίζουμε την 308 χωρίς την προφορική τροπολογία. Προσοχή. Ψηφίζουμε την 308 του κυρίου Γκρός χωρίς την προφορική τροπολογία. Το επαναλαμβάνω για να το αντιληφθούμε όλοι. διότι η συγκίτρια δεν δέχεται την ε, προφορική τροπολογία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 308 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της 308. Ποιος είναι κατά. Ω, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. ένας είναι αναποφάσιστος. Παραμένει αναποφάσιστος, πέρα της ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, γίνεται δεκτή η τροπολογία. Στη συνέχεια, τροπολογία 317 του κυρίου Φέρμπερ, υπέρ. κατά στο ΕΛΚ ε, πονάει το χέρι σας, γι' αυτό απέχετε τόσο πολύ. Τι συμβαίνει, την 317 του κυρίου Φέρμπερ, ποιος είναι υπέρ. Βλέπω ότι έχετε κουραστεί όλοι. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός παρακαλώ. Ψηφίζουμε την 317 άρχεται η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.16 και 3.36. Τις ψηφίζουμε μαζί. Κυρίου Φέρμπερ και κυρίας Μάισνερ. Ποιος είναι υπέρ αυτών των δύο. Κατά. Απορρίπτονται. 269-268. Οι τροπολογίες αυτές αποσύρονται. 340 και 313. Θα τις ψηφίσουμε μαζί γιατί είναι ίδιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Τρία δεκαπέντε. Του κυρίου Φέρμπερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 307 του κυρίου Κοχ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 302 του κυρίου Τσίλε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 304 του κυρίου Τσίλε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 342 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ με την προφορική τροπολογία υπαριθμών 4, τεχνικής φύσεως. Ή χωρίς, λέει ο πρόεδρος. Χωρίς την προφορική τροπολογία προφανώς, γιατί έτσι ζητήθηκε. Ψηφίζουμε την 342 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ χωρίς την τεχνική προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 341 καταπίπτει. Φτάνουμε στη 342 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ χωρίς προφορική τροπολογία, αλλά αυτό το ψηφίσαμε ήδη. 342 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και εάν δεν απατώμε φτάνουμε κατευθείαν στην 328. 321, 320, 19, 18, 297, 298, 299 ε, και 321. Τις ψηφίζουμε όλες αυτές μαζί, en bloc. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε για τις ηλεκτρονικής οδού. Πιστεύω ότι απορρίπτονται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται όντως. Και με μεγάλη πλειοψηφία. Η 301 αποσύρεται. Η 328 τώρα, του κυρίου Φέρμπερ. Τίθεται προς ψήφιση ακόμα. Ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλώς, την ψηφίζουμε λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της 328 του κυρίου Φέρμπερ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 322, 331 είναι ίδιες των κυρίων Ουλμερ, Βάισγερμπερ και Βίνκλερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Επομένως, Τώρα φτάνουμε αισίως στην 329. Ψηφίζουμε μαζί την 329, 323, 324, 325 και 326 γιατί είναι ίδια. Τις ψηφίζουμε on block. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε για τις ηλεκτρονικής οδού Νομίζω ότι απορρίπτονται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, κάποιος πάντοτε δεν ψηφίζει στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Και με μεγάλη πλειοψηφία. 27 κατά 13 ψήφοι υπέρ η 330 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε μόνο το σημείο Β. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 342 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία της κυρίας Τιτσάου. 303. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 337 του κυρίου Γκρός, Χωρί χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306. Ψηφοφορία κατά τμήματα είχε ζητηθεί εκ των προτέρων. Επομένως έτσι θα γίνει. Έχει κατατεθεί το έτοιμο αυτό. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της ε, τροπολογίας υπαριθμών 306 του κυρίου Κόχ. Από τη λέξη οχήματα μέχρι τη λέξη που παραδίδουν ε, ε, αντικείμενα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθέσουμε για της ηλεκτρονικής οδού, αν έχετε την καλοσύνη, ψηφίζουμε ηλεκτρονικό στο πρώτο τμήμα της 306. Κάντε μια προσπάθεια, ψηφίστε ηλεκτρονικά, δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 18 κατά. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 306. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Φτάνουμε λοιπόν εσίως στην 335 του κυρίου Κάστλερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φτάνουμε 305-338 των κυρίων Φέρμπερ, Βίσκερμπερ και Βίνκλερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτονται. 3.34 και 3.10 των κυρίων Κοχ και Μάισνερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 339 του κυρίου Κοχ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 332. Υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχει θέση. 332 του κυρίου Πίρκερ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Την 332 του κυρίου Πίρκερ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάποιος έχει ξεχάσει την ε, κάρτα ψηφοφορίας του. Πέρα της ψηφοφορίας, εν πάση περιπτώσει 22 υπέρ 19 κατά, εγκρίνεται. 3.14 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Η 105 καταπίπτει κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα ψηφίζουμε κάποιες τροπολογίες που έχουμε βάλει σε μία ομάδα. Τροπολογία 130. Σχεδόν στην τελευταία τελευταία σελίδα. Όλες οι υπόλοιπες ε, καταπίπτουν ή έχουν αποσυρθεί. Ως προσθήκη στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμό 17. Δεν υπάρχει δηλαδή αντίφαση. Κύριε Γκρόσο. Ναι. Αν κατάλαβα καλά την αιτιολογική σκέψη υπαριθμό 4, οι τροπολογίες καταπίπτουν αν η συμβαστική τροπολογία υπ. 21 γίνει δεκτή. Ε, αν έχει απορριφθεί το 321. Καλώς, ορθώς το έχω καταλάβει. Ναι, είναι δύσκολο γιατί είναι πολλές σελίδες το κείμενο και οι παραπομπές ε, αναφέρονται σε σελίδες πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους. Λοιπόν, ψηφίζουμε την προσθήκη της ε, συμβαστικής τροπολογίας υπαριθμών 17. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 του κυρίου Πίρκερ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 6 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 131 του κυρίου Τσίλε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 του κυρίου Κόχ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 του κυρίου Κόχ πάλι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 της κυρίας Τιτσάου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Ψηφίζουμε λοιπόν τελικά Ψηφίζεται λοιπόν τώρα για πρώτη φορά για την ομοθετική αυτή πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί. Πέρας της ψηφοφορίας, 28 υπέρ, 3 κατά. Δεύτερη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν για δεύτερη φορά για το νομοθετικό ψήφισμα αυτό. Αποσύρατε τις κάρτες σας. Δεύτερη ψηφοφορία παρακαλώ για άλλη μια φορά. Λυπάμαι, αλλά γίνονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, καθίστε σας παρακαλώ. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 110 του κυρίου Πίρκερ, η οποία θα κατέπιπτε εάν είχε εγκριθεί η 321. Παρακαλώ. Προτείνω λοιπόν σας αφήνω λίγο χρόνο να δείτε την τροπολογία 110 του κυρίου Πίρκερ. Είναι στη σελίδα 23 του εγγράφου που έχετε μπροστά σας. Θα το ξαναψηφίσουμε και βεβαίως θα ψηφίσουμε και τελικά το όλο κείμενο. Ψηφίζουμε την 110 του κυρίου Πίρκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε το κείμενο τελικά πρώτη ψήφιση της νομοθετικής πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία και ζητώ συγγνώμη γιατί ψηφίσαμε πριν χωρίς να έχουμε ψηφίσει την 110. Συνολική λοιπόν ψηφοφορία για αυτό το νομοθετικό ψήφισμα. Κάποιος δεν ψήφισε. Μία ψήφος λείπει. Κάποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται το ψήφισμα 25 υπέρ, 3 κατά 12 αποχές. Και δεύτερη ε, ψήφιση της νομοθετικής πρότασης, του νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεν είναι το ίδιο σκόρο. Όπως βλέπετε τώρα έχουμε 24 υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές. Το σημειώνουμε λοιπόν. Περιμένετε. Ε, πριν φύγετε παρακαλώ ε, τα διάφορα. Κάτι από τα διάφορα. Παρακαλώ. Περιμένετε λίγο. Μόνο ποιος έχει προστάτη ε, του επιτρέπω να σηκωθεί και να αποχωρήσει γρήγορα. Η κυρία Τιτσάου θέλει να προσθέσει κάτι. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Αντινούμπρα, consilierilor din uh, cadrul grupurilor politice pentru munca intensă pe care am desfășurat-o. Au fost câteva săptămâni în care am avut... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για την πολύ εντατική δουλειά ε, που κατέβαλαν. Επί σειρά ημερών ε, δουλέψαμε όλοι από κοινού επί ώρες. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία της Επιτροπής και την κυρία Ραμίνα Σπινέλη. Και Βεβαίως υποστηρίζω ότι το κείμενο μπορεί ακόμα να βελτιωθεί από σήμερα μέχρι την ε, ψήφιση στην Ολομέλεια και μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού μέσα στις προθεσμίες. Και είναι ένα πολύ καλό μήνυμα το οποίο διαβιβάζουμε στο Συμβούλιο ότι Ε, ε, ε, θα έπρεπε να λάβει υπόψη και την προηγούμενη Προεδρία, τις θέσεις της προηγούμενης Προεδρίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάναμε εμείς εδώ και στέλνουμε στην Ολομέλεια ένα πολύ καλό κείμενο. Λοιπόν, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα στο σημείο διάφορα. Το σημείο 15. Προσεχή συνεδρίαση 18 Ιουνίου από τις 15 έως τις 18 και 30 και στις 19 Ιουνίου από 9 έως 12 και 30 και 15 έως 18 και 30 πέρα τη συνεδρίαση. Γεια σας.